μέχρι 2 και 3 έως 5 το απόγευμα. Έχουν Δημιουργηθεί τα έγγραφα τη μέρη διάταξη. Είναι στα θέση σα μέσα από το ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα εύχομαι